ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό συμπέρασμα που μπορεί να συναγάγουμε από την απόψινή συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Αλμούνια. Εδώ κλείνει η συζήτηση για αυτή την προφορική ερώτηση. Έχουμε τώρα στην ημερήσια διάταξη τη δήλωση της Επιτροπής για τις Ευρωπαϊκές Δράσεις για τα θύματα της τρομοκρατίας. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Μπαρό, ο οποίος βρίσκεται ε, καθοδόν. Bonjour, monsieur le commissaire. Καλώς ήρθατε κύριε Επίτροπε. Έχετε το λόγο. Για πέντε λεπτά. J'associe à ces propos mon ami Joachim θύματα της τρομοκρατίας ε, είναι θύματα πράξεων εναντίον των δημοκρατικών αρχών των κοινωνιών μας. Αυτά τα θύματα αντιπροσωπεύουν την ανθρώπινη τραγωδία που είναι η τρομοκρατία. Και έχουμε προς αυτά τα θύματα ένα, μια υποχρέωση αλληλεγγύης, αναγνώρισης και υποστήριξης. Ο ρόλος της ε, Κομισιόν σε αυτόν τον τομέα είναι διτός. Πρώτον, θα πρέπει να βοηθήσει να εξασφαλίσει την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε ό,τι αφορά την κατάσταση και τα δεινά που ζουν τα θύματα της τρομοκρατίας. Και επίσης να ε, ενισχύσει την αντιπροσώπευση των συμφερόντων του σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εργαστεί προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω θύματα. Προκειμένου να εκριζωθεί η τρομοκρατία. Πρόκειται για την πολιτική πρόληψης. Από το 2004 και μετά η Κομισιόν υποστηρίζει οικονομικά ένα αριθμό σχεδίων που υλοποιούνται με στόχο να ενισχυθούν τα θύματα και οι τους μέσω κοινωνικής ή ψυχολογική υποστήριξη ε, μέσω οικονομικής ή ψυχολογικής υποστήριξης που χρειάζονται. Αυτά τα ε, σχέδια έχουν ως ε, κατεύθυνση την αύξηση της αλληλεγγύης που πρέπει να δειχθεί προς τα θύματα της τρομοκρατίας. Για το 2008 και μόνο, ο προπολογισμός των 2.200.000 ευρώ κατευθύνθηκε προς αυτή την προσπάθεια. Επιπλέον αυτών των δράσεων η Κομισιόν από το 2008 έχει δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο ενώσεων θυμάτων της τρομοκρατίας που έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την διακρατική συνεργασία ανάμεσα σε αυτές τις ενώσεις, αυτά τα σωματεία και να βελτιώσει την προάσπιση των συμφερόντων τους ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο προπολογισμό για αυτή τη δράση είναι 200.000 ευρώ. Αυτό το δίκτυο εργάζεται προς ε, πλήρωνες κατευθύνσεις. Αξιολογεί τις ενισχύσεις που δίδονται και την προστασία που χορηγείται σε αυτά τα θύματα σήμερα καθώς επίσης και ε, ενθαρρύνοντας, προωθώντας δραστηριότητες ε, για την διάδοση των βέλτιστων πρακτικών. Οι δραστηριότητες του δικτύου αποτελούν πολύ καλή βάση για τις δικές μας εργασίες στην Κομισιόν. Τέλος, Δεδομένου ότι η προστασία του πολίτη θα πρέπει να παραμένει πάντοτε στο κέντρο των πολιτικών μας, η Κομισιόν επιθυμεί στο μέλλον να ενισχύσει τη δράση τη στον τομέα της προστασίας των θυμάτων. Έχει σκοπό να υποστηρίξει, τα, να υποστηρίξει μέτρα που θα έχουν ως στόχο να ενθαρρυνθεί, να ενθαρρυνθεί θουν τα θύματα της ε, τρομοκρατίας ε, να καταθέτουν τις ματηρίες τους. Θέλουμε να ευαισθητοποιηθεί το κοινό, να προληφθεί η τρομοκρατία, γιατί μην ξεχνάμε ότι η τρομοκρατία πολλές, ε, η τρομοκρατία πολλές φορές αποτελεί καρπό ε, της, μιας, ενός φανατισμού και μιας πόλωσης. Και τέλος, ε, θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ειρήνης και προώθηση των δημοκρατικών αρχών. Η Κομισιόν λοιπόν έχει ως στόχο να ε, υιοθετηθεί μια χάρτα των δικαιωμάτων των θυμάτων της δημοκρατίας. Αυτά είχα να σας πω και σίγουρα προσωπικά συμμερίζομαι την αγανάκτησή την αγανάκτηση όλων που προκαλείται από τις ε, τρομοκρατικές δράσεις, ε, από τις τρομοκρατικές ανέργειες. Ε, θα πρέπει να δείξουμε την αλληλεγγύη μας στα θύματα της τρομοκρατίας. Αυτά κυρία Πρόεδρε. Θα ακούσω τις παρεμβάσεις των βουλευτών, των ευρωβουλευτών και θα απαντήσω. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ο λόγος στην κυρία Τερέσα Χιμένεθ Μπεθερίλ Μπάριο. Eh, eh, Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. οι περισσότεροι κυβερνώντες και πολίτες ε, θυμούνται τα θύματα της τρομοκρατίας μόνον αμέσως μετά από μια σημαντική τρομοκρατική πράξη όπως της Μαδρίτης, της Νέας Υόρκης, του Λονδίνου. Όταν ε, περάσει η πρώτη εντύπωση τείνουν να ξεχνούν και την απειλή της τρομοκρατίας και τα δικαιώματα των θυμάτων. Παρόλο ότι ε, δεν αμφισβητείται ότι η, η Κομισιόν είναι προσιλωμένη. έχει δείξει μια προσήλωση στην προάσπιση των δικαιωμάτων των αυτών. Για παράδειγμα στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης ε, που πρόσφατα ε, υιοθετήθηκε και αναγνωρίζεται ο ρόλος των θυμάτων και η σημασία της προάσπισης των δικαιωμάτων τους. Ε, η, η καταπολέμηση τρομοκρατίας πάντοτε βασιζόταν στην συνεργασία και στην, μεταξύ των κρατών και στην αλληλοεμπιστοσύνη, στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Αναρωτιέμαι όμως δεν θα ήταν καλό η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει μια Τη της νομοθεσίας των κρατών μελών σε ό,τι αφορά το θέμα των δικαιωμάτων των θυμάτων της τρομοκρατίας. Ε, η υιοθέτηση μιας Ευρωπαϊκής ε, Χάρτας Δικαιωμάτων των ε, Θυμάτων της Τρομοκρατίας θα ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα που θα βοηθούσε αυτούς που καταπολούν την τρομοκρατία και θα αποτελούσε κόλαφο για αυτούς που υποστηρίζουν την τρομοκρατία διότι τα θύματα με τη γενναιότητά τους και με την αξιοπρέπειά τους αντιπροσωπεύουν την αποτυχία της τρομοκρατίας και σίγουρα αντιπροσωπεύουν ταυτόχρονα ταυτόχρονα το μεγάλο θρίαμβο της δημοκρατίας. Μην ξεχνάμε ποτέ ότι το μόνο όπλο που έχουν οι αθώοι ε, ενάντια στην δημοκρατία είναι ο λόγος τους και η αναγνώριση της κοινωνίας. Συνεπώς, ας μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι ε, κανένας μας δεν βρίσκεται στο, απειρόβλητο. στο απειρόβλητο. Όλοι μπορούν να αποτελέσουμε θύματα της τρομοκρατίας. Οπότε η ερώτησή μου είναι η εξής θα συμφωνούσε η Κομισιόν να υιοθετηθεί μια Ευρωπαϊκή Χάρτα που θα αναγνωρίζει την, ε, ε, τα δικαιώματα των θυμάτων της δημοκρατίας και θα τα προωθεί και αν ναι, ποια μέτρα σκοπεύει να πάρει η καινούρια Κομισιόν για να προωθήσει ε, την σύνταξη μιας τέτοιας χάρτας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επιτροπέ για τα λόγια με τα οποία εκφράσατε την προσήλωσή σας μετά την ε, ε, της συνθήκης της Λισαβόνας ε, πλέον ε, το θέμα εμπίπτει στις της Κομισιόν. Ε, το πρόγραμμα της ε, Στοκχόλμης ε, πράγματι ε, περιλαμβάνει στο πολιετές 2009-2014 μια αναφορά στην αξιοπρέπεια των θυμάτων της τρομοκρατίας στα δεινά που έχουν ζήσει και στον ιδιαίτερα ευάλωτο χαρακτήρα τους αλλά πιο πολύ υπογραμμίζει το πρόγραμμα της Στοκχόλμης την ανάγκη προστασίας τους. Η Ισπανία θα αναλάβει την Προεδρία το επόμενο εξάμεινο, την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γνωρίζετε την αποφασιστικότητα της Ισπανίας στην καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας και όταν μιλώ για την Ισπανία εννοώ και την κυβέρνηση και την ε, κοινωνία. Ε, είμαστε αποφασισμένοι να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία σε όλες τις, τις μορφές. Συνεπώς θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε αυτή την εναρμόνιση, αυτό το πρόγραμμα πλαίσιο προστασίας των δικαιωμάτων των θυμάτων της δημοκρατίας στο πρόγραμμα δράσης που θα πρέπει να συντάξει η Ισπανική ε, κυβέρνηση για τα επόμενα χρόνια ε, και τα οποία, το οποίο πρόγραμμα δράσης θα μπορούσαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν το Βέλιο και η Ουγγαρία ως οι χώρες που θα αναλάβουν την Προεδρία ε, κατόπιν. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να επιβεβαιώσει το Κοινοβούλιο ε, την προσήλωσή του ε, και να ε, προωθηθεί και να προωθήσει μέσω του προγράμματος της Στοκχόλμης και μέσω της ε, νομοθετικής ατζέντα των επόμενων χρόνων ε, την αναγνώριση αυτών των δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την εναρμόνιση των, της προστασίας των δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Ο λόγος στην κυρία Μπιλμπάου Μπαραντίκα. Ε, ε, σύμφωνα με την τροπολογία που υπέβαλε η, Επιτροπή των Γυναικών υιοθετήθηκε, συμπεριλήφθηκε στην, ε, στο πρόγραμμα της Στοκόλμης και αυτό το θέμα, δεν υπήρχε στην αρχή. Έχουμε μάθει, εγώ προσωπικά έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα για την αξιοπρέπεια δουλεύοντας με τα θύματα της τρομοκρατίας τα τελευταία χρόνια και γι' αυτό το λόγο πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ενίσχυσης και αναγνώρισης των δικαιωμάτων δικαιωμάτων τους μέσω της πρώτον της αναγνώρισης των δεινών που, που έχουν ε, υποστεί ε, και τα θύματα είναι αυτοί που έχουν πληγεί άμεσα αλλά και οι οικογένειές τους. Ε, δεύτερον, θα πρέπει με υλικά μέσα να αποζημιώνονται και να προωθείται η μνήμη τους. Τρίτον, να εξανθρωπιστεί η συζήτηση για τα θύματα. Ε, τα θύματα υποφέρουν, θα πρέπει να τα προστατεύσουμε και θα πρέπει να τα βοηθήσουμε να τα συνδράμουμε. Θα πρέπει να μάθουμε μέσω της πολιτικής να μπαίνουμε μέσα στις καρδιές τους και, και, να εξανθρωπιστούμε. Τέταρτον, ε, δεν θα πρέπει η τρομοκρατία να χρησιμοποιείται ως πολιτικό όπλο. Ε, ασφαλώς έχουν υπάρξει τρομοκρατικές δράσεις ε, στην Ευρώπη, αλλά υπάρχουν και κυβερνήσεις οι οποίες έχουν ε, συμμετάσχει και έχουν εμπλακεί σε τέτοιου είδους ε, δράσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως η τρομοκρατία πλήττει την, τις ελευθερίες μας. Αφιερώνω αυτή μου την παρέμβαση στα θύματα της τρομοκρατίας. Ο λόγος κύριου κύριο Αγκουστίν μέρα. Το πρόγραμμα της Στοκόλμης περιλαμβάνει την εξή αναφορά, μεταξύ άλλων, υπέρ των θυμάτων της τρομοκρατίας. Τα θύματα της τρομοκρατίας χρειάζονται επίσης ιδιαίτερη προσοχή και ενίσχυση καθώς επίσης και κοινωνική αναγνώριση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δώσει αυτή την ενίσχυση και θα πρέπει να εξασφαλίσει την αναγνώριση εκ μέρους όλης της κοινωνίας σε όσους έχουν υποστεί την βαρβαρότητα της τρομοκρατίας. Θα πρέπει να αυτά τα άτομα να αποτελέσουν ηθική αναφορά. Και γι' αυτό το λόγο η προστασία του και η προστασία των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να ενισχύσουμε του πόρου οι οποίοι ε, χορηγούνται για την ε, ενίσχυσή του όπως ακριβώς το πρότεινε το, το ΕΛΚ μέσω της, ε, των τροπολογιών που υποβάλαμε στον προπολογισμό του 2010. Ανισχύθηκαν οι ενισχύσεις ε, κατά ένα εκατομμύριο ευρώ ε, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν σχέδια βοήθειας των θυμάτων και των οικογενειών τους μέσω η χρηματικής ή ψυχολογικής βοήθειας και επίσης για την χρηματοδότηση δικτύων και σχεδίων που έχουν ως στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινή γνώμης. Ένα τμήμα των πόρων ε, θα χρησιμοποιηθεί για την βελτίωση της δικαστικής συνδρομής των θυμάτων και των οικογενειών τους. Ένα στοιχείο. Η τρομοκρατία ίσων θύματα. Ε, τα συνολικά ποσά για την προετοιμασία και την πρόληψη τρομοκρατικών ενεργειών το 2000 ε, 10 θα φτάσει στα 21.300.000 ευρώ. Η Τερέσα ε, ε, ε, έχει ως στόχο στις προτάσεις της να γίνουν πιο ορατά τα θύματα και εμείς θα πρέπει να βοηθήσουμε. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε με μια γραπτή δήλωση, μετά με ένα ψήφι, να συνεχίσουμε με ένα ψήφισμα και στο τέλος να καταλήξουμε σε ένα πολιτικό ψήφισμα όλων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες μας. Τα θύματα μας ε, δημιουργούν αισθήματα αλληλεγγύης, συμπόνιας, αναγνώρισης, αξιοπρέπειας. Ε, μας δημιουργούν αναμνήσεις ε, και αντιπροσωπεύουν την καταπάτηση όλων των αρχών της δικαιοσύνης. Ευχαριστώ πολύ. Merci beaucoup. Ε, et Κύριε Βαρό, δεν ε, ε, ε, είναι, δεν τυχαίο που όλοι οι μιλητές είναι Ισπανοί σήμερα. Εκτός από την τρομοκρατία, τα θύματα στη χώρα των Βάσκων υφίστανται πολύ συχνά την σιωπή ή την περιφρόνηση. Και τα θύματα, γι' αυτό το λόγο, απαιτούν μια πολιτική που θα τα αφορά. Ε, θα ήθελα να προσθέσω δύο λόγια στα όσα είπαν οι προηγούμενοι ομιλητέ. Υπέρ μιας χάρτας ε, ε, ή μιας σύγκλησης των δρασιών μας με δέκα σημεία. Πρώτον, η πολιτική των θυμάτων απαιτεί μια δημόσια συνοδεία, αναγνώριση, κοινωνική αναγνώριση των θυμάτων. Δεύτερον, γρήγορη και αποτελεσματική αποζημίωση των ζημιών. Τρίτον, ίση μεταχείριση σε όλα τα θύματα. Τέταρτον, μια πολιτική συνένεση, πολιτική και κοινωνική συνένεση για τα μέτρα που είναι απαραίτητα υπέρ των θυμάτων της τρομοκρατίας. Πέμπτον, πολιτική ε, καταδίκης των, ε, της βίας. Έκτον, υποδειγματική ε, τιμωρία των, ε, των υπετίων. Έβδομον, μια διδακτική, μια παιδαγωγική κατά της βίας ε, προς τον πληθυσμό. Ε, εγγύηση ε, μη επανάληψης που θα πρέπει να δίδεται στα θύματα. Ένατον, πολιτική διατήρηση της μνήμης για να αποφύγουμε την ιστορική λύθη. Και δέκατον, μια πολιτική ε, κοινωνική συμφιλίωσης για να θεραπευθούν οι πληγέ της τρομοκρατίας. Αυτά είναι τα δέκα σημεία τα οποία προτείνω ως κεντρικά για μια πολιτική υπέρ των θυμάτων της τρομοκρατίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Έχουν ζητήσει τρεις ομιλητές το λόγο. καταρχά, ο κύριος Παπα-Νικολάου οι επιθέσεις σε μαδρίτη και λονδίνο αλλά και τα πρόσφατα χτυπήματα στη δική μου χώρα στην ελλάδα καταδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος της τρομοκρατίας. η τρομοκρατία απειλεί τον τρόπο ζωής και την ελευθερία μας. δεν στοχοποιεί μόνο τα άμεσα θύματα ή τις οικογένειές τους οι οποίες επίσης άμεσα πλήττονται αλλά ολόκληρη την κοινωνία. τα ευρωπαϊκά πιλωτικά προγράμματα που αναφέρθηκαν για τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων είναι ένα θετικό δείγμα για την ανακούφιση των πληγών ωστόσο μένουν πολλά ακόμα να γίνουν η βοήθεια των θυμάτων και των οικογενειών τους δεν είναι μόνο ηθικά επιβεβλημένη είναι κυρίως επιβεβλημένη ώστε να στείλουμε στην τρομοκρατία ένα καθαρό μήνυμα ότι δεν ξεχνάμε. δεν ξεχνάμε αποτρόπαιες πράξεις που στιγματίζουν τη δημοκρατία και τη συνοχή μας. δεν ξεχνάμε ότι θύματα της τρομοκρατίας είναι συχνά ανυποψίαστοι πολίτες που τραυματίζονται ή σκοτώνονται ενώ εκτελούν τις καθημερινές τους ασχολίες δεν ξεχνάμε ότι στην ευρώπη που δίδαξε την ανοχή και τη δημοκρατία οι πράξεις βίας δεν θα είναι ποτέ ευπρόσδεκτες. σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ε, υποστηρίξω την πρόταση της κυρίας Τζιμενέλ Τετσερίμ σχετικά με ένα ε, ευρωπαϊκό χάρτη για τα ε, θύματα και τις οικογένειες των θυμάτων της τρομοκρατίας και να υπογραμμίσω ότι εδώ έχουμε μια καταπληκτική ευκαιρία υπάρχει μια καταπληκτική ευκαιρία για την Ευρώπη να δώσει μια διαφυζήτητη ένδειξη όσον αφορά την έννοια της τρομοκρατίας λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία ε, μιας τέτοιας στάσης προκάλεσε το 2005 την ε, ε, χρεοκοπία της διαδικασίας της Βαρκελόνης όταν οι αρχηγοί των κρατών και κυβερνήσεων των ευρωμεσογειακών χωρών δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν και έτσι λοιπόν σήμερα έχουμε μια εξαιρετική ευκαιρία για να ξαναξεκινήσουμε σε νέα βάση τον διάλογο με την άλλη όχθη της Μεσογείου ε, με βάση μια σαφή διακήρυξη όσον αφορά την έννοια που απαιτεί τη βάση του πολιτισμού μας και του ανθρωπισμού μας δηλαδή που είναι το ιερό της ιερότητα της ζωής. Ευχαριστώ και τέλος η κυρία Ντότς. Thank you, Madam President. Ευχαριστώ κυρία ε, και κύριε Μπαρό. Ε, κύριε Επίτροπε, είμαστε ευγνώμονε για την υποστήριξή σας για τα θύματα της τρομοκρατίας. Αυτό είναι και σωστό και δίκαιο. Και βεβαίω αναγνωρίζουμε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα στη Βόρεια Ιρλανδία μέσω του ειρνευτικού προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε εκεί. Θα πρέπει να ξέρει η Κομισιόν ότι η Βόρεια Ιρλανδία αντιμετωπίζει εκ νέου ε, νέα τρομοκρατική απειλή από ρεπουμπλικάνικες ε, οργανώσεις και η κατάσταση είναι κρίσιμη στη Βόρεια Ιρλανδία. Η Διεθνή Επιτροπή Παρακολούθηση ε, πέστησε την προσοχή σε πρόσφατε επιθέσει. Δύο στρατιώτε που ετοιμάζονταν να, πάνε για, να φύγουν για το Αφγανιστάν ε, ε σκοτώθηκαν, καθώ επίση και ένα αστυνομικό. Η Κομισιόν ε, προσδιορίζει τους βασικούς στόχους να κοινοποιηθεί το κοινό εναντίον της τρομοκρατίας σε όλες τις μορφές. Παρ' όλα αυτά όμως θεωρώ ότι με τη μετάβαση στο ευρύτερο πρόγραμμα ε, ειρήνευσης ε, χάθηκε αυτός ο στόχος. Καλωσορίζω ε, την ύπαρξη μιας Ευρωπαϊκής Χάρτας για τα θύματα και θα ήθελα να γίνει μια σαφή διαφοροποίηση ανάμεσα στα θύματα της τρομοκρατίας και τους ε, δράστες τρομοκρατικών ε, ενεργειών. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Γκάδενμπακ. Ευχαριστώ ω Αυστριακή εδώ και πολλά χρόνια δόξα τω Θεώ, δεν είχαμε τρομοκρατικά χτυπήματα. Θα ήθελα να προσθέσω να συμφωνήσω με τον συνάδελφο, γιατί ναι μεν χρειαζόμαστε αφενός την υποστήριξη των θυμάτων, αλλά αυτό που παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει είναι ο βιότοπος εκείνος, ο οποίος θα αποξηράνει, αν θέλετε, τις επιθέσεις της τρομοκρατίας. Θα πρέπει λοιπόν εμείς ως Ευρωκοινοβούλιο να χρησιμοποιήσουμε σκληρή γλώσσα. Και νομίζω ότι πάντα μιλάμε για ανοχή, αλλά σε έναν τομέα δεν επιτρέπεται η ανοχή εκεί όπου χρησιμοποιείται βία. Ευχαριστώ. Ε, παρεμβάσεις αυτές που είναι τόσο φορτωμένες με ε, αξιοπρέπεια αλλά και αγανάκτηση ε, και σας ευχαριστώ εκ μέρους ε, της Προεδρίας για, όλους, για όλες τις παρεμβάσεις. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Παρό. Κυρία Πρόεδρε, πολύ σωστά υπογραμμίσατε πως η συζήτηση αυτή ήταν φορτωμένη, με, φορτωμένη συγκινησιακά. Όλοι μας αυτή τη στιγμή σκεπτόμαστε τα θύματα ε, που έπεσαν κάτω από τα χτυπήματα της τρομοκρατίας με τρόπο πραγματικά ε, τυφλό και άδικο. Όπως το είπε ο κύριος Λόπες Αγκουίλα, είναι μια τρομερή μορφή εγκληματικότητας. Αυτό που ήθελα να σας πω λοιπόν είναι ότι πρώτα απ' όλα το πρόγραμμα της Στοχόλμης πραγματικά αξιοποιεί τονίζει μάλλον την ε, μοίρα των θυμάτων. Υπάρχει μια ευρωπαϊκή πολιτική δέσμευση να δώσουμε πολύ περισσότερη προσοχή στα θύματα του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Ε, θα έπρεπε να πω στην κυρία Τερέζα Μπεσερίλ ότι πράγματι θα κατευθυνθούμε προς ε, ένα χάρτη των δικαιωμάτων των θυμάτων της τρομοκρατίας. Όπως πολύ, πολύ καθαρά το διατύπωσε η κυρία με ε, την ε, πολύ οδυνηρή προσωπική εμπειρία που έχει ε, του θέματος αυτού. Επίσης πιστεύω ότι θα αναλύσουμε το 2010 όλες τις ελλείψεις που υπάρχουν σήμερα όσον αφορά την προστασία των θυμάτων της τρομοκρατίας στα διάφορα κράτη-μέλη. Πράγματι έχετε δίκιο ότι με τον ΑΒ τρόπο πρέπει να καταφέρουμε να εναρμονίσουμε την νομοθεσία μας ε, όσον αφορά την τρομοκρατία και τα θύματα της τρομοκρατίας. Πρέπει πραγματικά η Ευρώπη να αντιδράσει ε, με μία ενιαία ε, κίνηση εναντίον της τρομοκρατίας. Και με βάση αυτή τη μελέτη θα δούμε πώς θα μπορέσουμε στην πράξη να εναρμονίσουμε και να προσεγγίσουμε όλα αυτά τα μέτρα που θα μπορέσουν να βελτιώσουν την κατάσταση των θυμάτων ε, της τρομοκρατίας στην Ευρώπη. Αυτό θα είναι το αντικείμενο του σχεδίου δράσης. Και είναι απολύτως βέβαιο ότι θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα της προστασίας των θυμάτων με βάση πράγματα που ελέγχθησαν κατά τη συζήτηση. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, ότι θα πρέπει πρώτα απ' όλα να κάνουμε γνωστό το δράμα και τα δεινά που υποφέρουν ε, τα θύματα της τρομοκρατίας που πολύ συνακαλύπτουν από σιωπή, αν όχι και από περιφρόνηση. Δεύτερον, πολύ σωστά πρέπει να υπάρχει ταχεία αποζημίωση των θυμάτων. Έχετε δίκιο που το τονίζετε αυτό. Ε, και επίσης αναφερθήκατε στο θέμα της απονομιμοποίησης του λόγου της τρομοκρατίας. Δεν μπορούμε να νομιμοποιούμε ένα λόγο που με τον ΑΒ τρόπο μπορεί να νομιμοποιεί την ιδέα του τραυματισμού ή της θανάτωσης ε, αθώων θυμάτων και ότι αυτό μπορεί να εξυπηρετεί με οποιοδήποτε τρόπο την ανθρωπότητα. Πρέπει πραγματικά να βάλουμε φρένο σε αυτή την ε, έκφραση ε, που ε, είναι εναντίον κάθε ε, αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, έχει χρηματοδοτηθεί με ένα εκατομμύριο ευρώ το πρόγραμμά μας για τη βοήθεια των θυμάτων. Ε, Πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που ο Ιωκή Αλμούνια βρίσκεται στο πλευρό μου σήμερα γιατί πρέπει να σας πω ότι και οι δυο ε, θα ε, δεσμευτούμε εκ μέρους της Κομισιόν και θα πιέσουμε ε, ούτως ώστε στα πλαίσια του προγράμματος της Οχόλμης η ε, Ευρώπη να αποκτήσει ένα υποδειγματικό πρόγραμμα για την ε, προστασία και την αρρωγή των θυμάτων της τρομοκρατίας. Αυτές είναι οι απαντήσεις που ήθελα να δώσω στις ερωτήσεις σας και να είστε σίγουροι ότι δεν είμαστε αδιάφοροι ούτε εγώ ούτε ο Κιμ Αλμούνια απέναντι σε αυτά που μας είπατε. Ευχαριστώ. Σας προτείνω ε, για να μην περάσουμε αμέσω στην επόμενη συζήτηση, να κρατήσουμε ενό λεπτού σιγή, σιωπής για όλα τα θύματα της τρομοκρατίας. Ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις, σας λοιπόν. Ε, τώρα στην ημερήσια διάταξη έχουμε ένα άλλο θέμα πιο τεχνικό αυτή τη φορά για ένα θέμα επικουρικότητας. Για να αρχίσουμε τη συζήτηση.